Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω θερμά στη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Να περιμένω λίγο μέχρι να βάλετε όλοι τα ακουστικά σας. Αποφάσισα να μιλώ στην μητρική μου γλώσσα από εδώ και πέρα αφού υπάρχει αυτή η πολυτέλεια και έχουμε καταπληκτικούς διερμηνείς, αποφάσισα να μιλήσω γερμανικά σήμερα. Αξιότιμοι βουλευτές, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, πριν δώσω το λόγο στον εξέχοντα προσκεκλημένο μας που είναι αρμόδιος από τη Φιλανδική Προεδρία για θέματα συνεργασία και ισότητα. Πριν δώσω λοιπόν το λόγο στον κ. Τόμα Μπλόμπκβιστ, θέλω να σα ρωτήσω αν έχετε κάποια αντίρρηση για τη μερίσια διάταξη. Συμφωνείτε και αν συμφωνείτε, προχωρούμε στο επόμενο σημείο τη μερίσια διάταξη, που είναι οι ανακοινώσει τη Προέδρου. Έχω να σα κάνω κάποιε ανακοινώσει 4 Σεπτεμβρίου. Το 2019 είχαμε μια συνεδρίαση και έπειτα σε γραπτή διαδικασία στις 10 Σεπτεμβρίου έχουν αποφασίσει οι συντονιστές τα εξή. Πρώτα απ' όλα να γίνει σύνταξη δύο νομοδοτήσεων σε ό,τι αφορά το ΕΚΙ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το οικονομικό έτος 2018 και την σύνταξη αυτή τη, ε, μάλλον αυτών των χρηματοδοτήσεων, θα αναλάβει η κυρία Φράνσις Φιτζέραλντα από την ομάδα του ΕΛΚ. Έπειτα αποφασίσαμε να γίνει ε, μια γραπτή νομοδότηση σε ό,τι αφορά την έκθεση της Επιτροπής για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ντρουά, σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό. Μιλάμε για τη χρονιά 2018. Και άλλη απόφαση, αποφασίσαμε, έλεγα, να συνεχίσουμε το έργο της προηγούμενης θητείας για δύο νομοθετικά ζητήματα που αφορούν τις γυναίκες στα Διοικητικά Συμβούλια και τη Συμφωνία της Κωνσταντινούπολης. Ε, θα είναι η πρόεδρος που η εισηγήτρια για το θέμα γυναίκες στα Διοικητικά Συμβούλια, δηλαδή την ισότητα των ε, φύλων. Ε, στα ΔΣ, ενώ την σύμβαση της Κωνσταντινούπολης θα την αναλάβει η ομάδα του ΕΛΚ. Και σύντομα θα μας ε, πούν ποια ή ε, ποιος είναι από τη δική τους πλευρά. Επίσης, αποφασίστηκε να υπάρξει και μία ομάδα εργασίας για το ΕΚΙ, στην οποία θα συμμετέχουν όλες οι ομάδες, δηλαδή το Ευρωπαϊκό το για την Ισότητα των Φύλων. Επίσης, η κυρία Φερακού και η κυρία Ζαχαροπρούλου, η μία ως μέλος και η δεύτερη ως αντικαταστάτρια θα είναι αρμόδιες ε, στο πλαίσιο του δικτύου για την εφαρμογή της Σύμβασης των Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Επίσης, ε, στο δίκτυο των αναφορών μέλος θα είναι η Οχένια Ροτρίγκες Παλόπα δεν έχει ακόμη οριστεί ο αναπληρωτής, ε, έχει αναβληθεί η διαδικασία αυτή μέχρι να έχουμε τις υποψηφιότητες. Επίσης, ε, ε, δόθη έγκριση για τη διεξαγωγή δύο ανοιχτών ακροάσεων στο πλαίσιο αυτής της χρονιάς. Η πρώτη θα λάβει χώρα 18 Νοεμβρίου στο πλαίσιο της Διεθνούς ημέρας για την καταπολέμηση της ασφάλειας των γυναικών και η δεύτερη ακρόαση αρχές Δεκεμβρίου με θέμα τη Στρατική τη Ένωση ε, για την ισότητα των φύλων 2020-2024. Βλέπετε ότι ήταν πολύ παραγωγική η συνεδρίαση των συντονιστών, είχαμε πολλά θέματα. Και τώρα, αν ε, συμφωνείτε, να περάσουμε στο επόμενο σημείο που είναι η έγκριση των πρακτικών της συνεδρίας 10 Ιουλίου. Αν δεν υπάρχουν ε, παρατηρήσεις, θεωρώ ότι εγκρίνεται και αυτό το σημείο. Και τώρα φτάνουμε στο ε, σημαντικό σημείο της μερισιάς διάταξης ε, ε, που έχουμε την παρουσία της Προεδρίας Συμβουλίου και συγκεκριμένα έχουμε προσκαλέσει σήμερα τον κύριο Τόμας Μπλόγκβιστ, Υπουργό για τη Σκανδιναβική Συνεργασία και την Ισότητα των Φίλων από την Φιλανδική Προεδρία και την ομάδα του. του. Σας καλωσορίζω. Ήδη ξέρω ότι είσαστε προχωρημένοι στην εργασία σας ήδη και στην Ολομέλεια ήδη ακούσαμε μια πάρα πολύ ε, εντυπωσιακή ομιλία της Μαθητικής Προεδρίας στο Στρασβούργο σε ό,τι αφορά την συνεργασία και την ε, ισότητα των φύλων που είναι προτεραιότητες. Είναι η ενδυνάμωση των κοινών μας αξιών και το κράτος δικαίου επίσης ε, σημαντικά ζητήματα, όπως και άλλο που αναφέρετε. για μας είναι προτεραιότητα. Θα ήθελα να σας δώσω το λόγο για 15 λεπτά περίπου, ώστε να μας παρουσιάσετε λίγο την κατάσταση και εν συνεχεία, όπως έγινε και την προηγούμενη φορά, θα δώσω το λόγο καταρχάς ε, στους συντονιστές και εν συνεχεία φυσικά οποιοδήποτε άλλο συνάδελφος μπορεί να συμπληρώσει με παρατηρήσεις, ερωτήσεις ή σχόλια στην παρουσίαση του κυρίου Μπλόμκβιστ. Καλώς ήρθατε εκ νέου λοιπόν κύριε Υπουργέ στη συνεδρίασή μας και παρακαλώ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση σε αυτή την πάρα πολύ σημαντική ε, σειρά συζητήσεων. Όπως και η Πρόεδρος, θα μιλήσω και εγώ τη μητρική μου γλώσσα για την εισαγωγή μου. Ε, κατά τη διάρκεια όμως της διαδικασίας των ερωταποκρίσεων μπορεί να απαντήσω και σε άλλη γλώσσα, να χρησιμοποιήσω και τα φιλανδικά, γιατί τώρα θα μιλήσω σουηδικά, που είναι η μητρική μου γλώσσα. Καταρχάς, θα ήθελα να τονίσω εξ ονόματος ε, της ε, Προεδρίας του Συμβουλίου ότι προσβλέπουμε σε επικοδομητική συνεργασία. Θα ήθελα να συγχαρώ την ε, Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους και όλα τα μέλη της Επιτροπής σας για τον διορισμό του στην Επιτροπή και θα ήθελα να συνεχιστεί η αγαστή συνεργασία στη διάρκεια της Φιλανδικής Προεδρίας αλλά και μετά την Προεδρία. Η Φιλανδική Προεδρία μπορώ να πω ότι δεσμεύεται ιδιαίτερα σε θέματα ισότητας των φύλων. Πρόκειται για κάτι το οποίο εντάσσεται στο κυβερνητικό μας πρόγραμμα υποστηρίζεται από υπουργούς και η σύνθεση της κυβέρνησης ε, περιλαμβάνει 11 γυναίκες υπουργούς. Υπάρχει ισχυρή δέσμευση για ίσες ευκαιρίες και ισότητα των φύλων. Η κυβερνητική μας πολιτική περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα για ίσες ευκαιρίες και την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών και επίσης ε, κάνουμε και μεγάλη προσπάθεια για να υπάρχει διαφάνεια στο θέμα των μισθών. Και θέλουμε να κάνουμε και αλλαγές στην νομοθεσία που θα αντανακλούν ακριβώς αυτό το στόχο. Υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι όσον αφορά την ισότητα των φύλων που σχετίζονται και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, προσβλέπουμε σε μια νέα στρατηγική για την ισότητα των φύλων και ε, δίνουμε και μάχη προκειμένου να υπάρχει ισότητα των φύλων και σε θέματα προπολογισμού. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα για μας. Αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίχους ε, πάνω στους οποίους θέλουμε να χτίσουμε την ε, πολιτική μας. Οι ίσες ευκαιρίες είναι ένας τρόπος να επιτευχθούν οι στόχοι του ε, τρίου των Προεδριών. Ε, η Ρουμανία και η Κροατία είναι οι άλλες δύο χώρες και ε, μαζί με αυτές θεωρούμε ότι το φιλανδικό κυβερνητικό πρόγραμμα αποτελεί καλό σημείο κίνησης για την επίτευξη αυτών των στόχων. Οι προτεραιότητές μας είναι να ενισχύσουμε τις κοινέ μας αξίες και η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει μια ένωση η οποία θα είναι πιο ανταγωνιστική και ε, θα περιλαμβάνει όλη την κοινωνία. Θέλουμε να είμαστε επίσης ε, ηγέτες σε θέματα ε, κλιματικών, κλιματικής αλλαγής και να ενισχύσουμε και την ασφάλεια. Όλες οι προτεραιότητές μας έχουν άμεση σχέση με την ανάπτυξη και της κοινωνικής διάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι προτεραιότητές μας επίσης σχετίζονται άμεσα με την ισότητα των φύλων που είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη προκειμένου να επιτευθούν οι άλλοι κεντρικοί στόχοι. Οι προτεραιότητές μας επίσης συνάδουν και με τις νέες ε, κατευθυντήριες γραμμές ε, της νέας πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η κυρία Βάντερ Λάιεν επισήμανε τις προτεραιότητες της, οι οποίες είναι ε, και οι προτεραιότητες οι οποίες υποστηρίζουμε και εμείς ακράδαντα και χαιρόμαστε που για πρώτη φορά υπάρχει γυναίκα πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρόκειται για μια πάρα πολύ θετική ένδειξη στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ισότητα των φύλων. Στη διάρκεια της Προεδρίας ε, θα επικεντρωθούμε στη στήριξη της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επόμενη πενταετία ε, και για το στρατηγικό σχεδιασμό. Επίσης, ε, κάνουμε προσπάθειες προκειμένου να υπάρχει συνέχεια και η μετάβαση ανάμεσα στις διάφορες ε, προεδρίες, ε, στα καθήκοντά τους ε, και στις αρμοδιότητές τους να γίνεται με πιο ομαλό τρόπο. Να προχωρήσουμε μαζί για καλύτερη οικοδόμηση της Ευρώπης, να βρούμε ένα καλύτερο τρόπο να προχωρήσουμε και να μπορούν και τα κράτη-μέλη, είτε μεγάλα είτε μικρά, βόρεια, νότια, ανατολικά ή δυτικά, να μπορούν να βιώσουν το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντική για αυτούς. Βεβαίως η ισότητα των φύλων είναι ένα απόσπαστο τμήμα όλων αυτών και εμείς ε, προσβλέπουμε σε μια βιώσιμη στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία στρατηγική θα μπορέσουμε να επιτύχουμε ισότητα των φύλων. Η, μια άλλη προτεραιότητα της Προεδρίας μας είναι η οικονομία της ευημερία της πρόνοιας. Αυτό θεωρούμε ότι θα επηρεάσει την ευρωπαϊκή στρατηγική για το μέλλον και θα αποτελήσει και ε, σημαντικό σταθμό για την ανάπτυξη της κοινωνικής διάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, η οικονομία της πρόνοιας σχετίζεται ε, άμεσα με τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Πυλώνα και εμείς υποστηρίζουμε την εφαρμογή αυτού του πυλώνα. Πρόκειται για κάτι το οποίο βοηθά την οικονομική ανάπτυξη, αλλά ταυτόχρονα με την ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης. Πρόκειται λοιπόν για δύο πυλώνες οι οποίες συνεργάζονται ε, και δεν είναι ο ένας αντίθετος στον άλλον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να μπορέσουμε να εντάξουμε και την διάσταση του φύλου στην οικονομική πολιτική και στη διαδικασία του προπολογισμού. Στόχος μας είναι να εντάξουμε περισσότερο τις πολιτικές για το φύλλο σε όλες τις ε, ευρωπαϊκές πολιτικές, ιδίως όσον αφορά τον προγραμματισμό μετά το 2020. Η ισότητα των φύλων είναι τμήμα της βιώσιμης ανάπτυξης. Δεν μπορούμε να επιτύχουμε τους στόχους μας για το 2030 χωρίς μια ισχυρή διάσταση του φύλου σε όλους τους τομείς πολιτικής. βάση αυτού έχουμε και τη διάσκεψη Ευρώπη για την ισότητα των φύλων στο Ελσίνκι την επόμενη εβδομάδα. Και εμείς υποστηρίζουμε και την κατεύθυνση ε, των ε, στόχων ε, των Ηνωμένων Εθνών. Η στόχη βιωσιμότητα των Ηνωμένων Εθνών είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε να εφαρμόσουμε εδώ και 20 χρόνια και θεωρούμε ότι θα πρέπει να δούμε και τι θα γίνει στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ την όλη διαδικασία και αυτό μας βοηθά να προετοιμάσουμε την πολιτική για τα φύλλα για την επόμενη πενταετία. Το η μελλοντική πολιτική για την ισότητα των φύλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτι ε, στο οποίο επικεντρώνεται η Φιλανδική Προεδρία και ο στόχος μας είναι το Δεκέμβριο το Συμβούλιο να εγκρίνει συμπεράσματα για το θέμα αυτό. Στην ίδια συνεδρίαση θα γίνει και μια συζήτηση πολιτικής για τη μελλοντική πολιτική για την ισότητα των φύλων με ιδιαίτερη εστίαση σε θέματα ολοκλήρωσης και ένταξης των δύο φύλων. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που αφορούν ε, ε, το φύλλο, στα οποία θα ήθελα να σταθώ. Θέλουμε να έχουμε μια ασφαλή και προστατευμένη Ευρώπη για όλους. Ε, το να πάψει να υπάρχει το χάσμα ε, μισθών μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι ένας πολύ σημαντικός στόχος και σίγουρα πρέπει να επιτευχθεί. Πρέπει επίσης ε, να υπάρχουν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού και μεταξύ κρατών μελών, ιδίως ε, όσον αφορά τον κοινωνικό πυλώνα και τις ε, αμοιβόμενες θέσεις εργασίας επί ίσης όρης, κάτι το οποίο προσπαθούμε να έχουμε. Αν ενισχύσουμε τους ίδιους μισθούς, θα μπορέσουμε να μειώσουμε και το χάσμα που υπάρχει στις συντάξεις. Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα είναι να καταπολεμήσουμε τη βία κατά των γυναικών και να προστατεύονται τα, θέματα, τα θύματα Ευτής εξ αρχή, ε, στο Συμβούλιο της Ευρώπης η Φιλανδία έχει μεγάλη υποστήριξη για την προώθηση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολη, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Θέλουμε λοιπόν να προωθήσουμε την κύρωση της Σύμβασης τη Κωνσταντινούπολη από όλα τα κράτη-μέλη και θέλουμε να ε, συμβάλλουμε έτσι και στην ένταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην σύμβαση αυτή. Επιπλέον, θα ήθελα να τονίσω και μία τάση η οποία είναι πάρα πολύ ψηλή και έχουμε να την αντιμετωπίσουμε για το μέλλον. Οι τεχνολογικές εξελίξεις, οι οποίες ε, φυσικά ε, συνοδεύονται και από πάρα πολλές ευκαιρίες ε, για την ανάπτυξη της αγοράς εργασίας και τον, την αλλαγή των συνθηκών εργασίας. Ταυτόχρονα όμως θα μπορούσαν να είναι και απειλή για τη θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας. Και αυτό φυσικά αποτελεί τεράστια πρόκληση. Υπάρχει υποεκπροσώπηση των γυναικών στον ψηφιακό και τεχνολογικό τομέα και πολύ συχνά οι γυναίκες είναι θύματα παρενόχλησης στο διαδίκτυο. Στη διάρκεια της ε, Φιλανδικής Προεδρίας προωθούμε νομοθεσία για τα θέματα αυτά για την προώθηση της ισότητας των φύλων. Υπάρχει το σχέδιο οδηγίας ε, για τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια ε, που στόχο έχει ε, να υπάρχει η ισότητα των φύλων στις επιχειρήσεις και φυσικά θέλουμε και μεγαλύτερη υποστήριξη για την νομοθετική αυτή πρόταση η πρόεδρος της Επιτροπής, η κυρία Βαντερ Λάιεν, ε, τόνισε ότι στόχος της είναι να συνεχίσει να υποστηρίζει τη συγκεκριμένη νομοθεσία και εμείς ε, θα συνεχίσουμε να την υποστηρίζουμε αν πληρούνται φυσικά οι προϋποθέσεις στο Συμβούλιο. Πρόκειται για μια οδηγία η οποία ήταν στα σκαριά εδώ και 10 χρόνια. Παρά τις προσπάθειες, ε, οι διαπραγματεύσεις ακόμα δεν έχουν καρποφορήσει στη διάρκεια της Φιλανδικής ε, Προεδρίας θα κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να πατάξουμε τις διακρίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα γίνει μια συζήτηση πολιτική τον Οκτώβριο με τους Υπουργούς Απασχόλησης, θα δούμε τα θέματα της διάκρισης και η μεγαλύτερη πρόκληση σε αυτή την περίπτωση είναι να βρούμε τον καλύτερο και πιο αποτελεσματικό τρόπο να βελτιωθεί η κατάσταση. Ο στόχος των συζητήσεων είναι να υποστηρίξουμε τη Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να συνεργαστούμε ε, και με τις ε, επόμενες προεδρίες. Αυτά όλα φυσικά μπορούμε να τα βασίσουμε στη συμβολή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, με την ισχυρή υποστήριξη και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Χαιρόμαστε που υπάρχει ήδη συμφωνία για την οδηγία για την ε, ισορροπία εργασιακού και οικογενειακού βίου, αλλά το επόμενο βήμα είναι η εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Η οδηγία αυτή θέλει να επιτύχει ισορροπία μεταξύ ανδρών και γυναικών, που είναι μία από τις βασικές προκλήσεις στο χώρο της εργασίας. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και περιμένω τις ε, σκέψεις, ε, τις αντιδράσεις σας και φυσικά θα κάνω ό,τι μπορώ για να απαντήσω σε τυχόν ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Υπουργέ. Ήταν μια περιεκτικότατη ε, παρουσίαση. Μετά από την δική σας λοιπόν ε, ομιλία και μετά και την ε, παρουσίαση του προγράμματος της Αναδικής Προεδρίας ε, είμαστε αισιόδοξοι με τις πολύ ωραίες εικόνες τις οποίες εσείς μας περιγράψατε. Θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα καταρχάς όπως είπα στους συντονιστές από το ΕΛΚ κυρία Νόχελ και μετά σε μοίρα Ραφαέλ. So the next. No. Uh, ah, Φαντάζομαι ακούτε και από εδώ και να ευχαριστήσω το γείτονα <laughs> κυρίως που ε, αλλάζει θέση μαζί μου για να μπορέσω να μιλήσω. Λοιπόν, ήθελα πρώτα απ' όλα και εγώ ε, να συμφωνήσω ε, με αυτό που είπε η Πρόεδρος και από την εισαγωγική σας παρέμβαση είπατε ότι και κάνατε σαφές ότι είναι πάρα πολύ προσιλές για σας το θέμα της ισότητας των φύλων. Έχετε αναφέρει πολλούς τομείς στους οποίους υπάρχει συμμετοχή γυναικών και πρέπει να δείτε ιδιαίτερη σημασία στις γυναίκες και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί αυτό που δεν θα θέλαμε θα ήταν μια προεδρία που θεωρεί ότι ένα θέμα υπάρχει, ένα θέμα είναι αυτό το οποίο θα την απασχολεί κυρίω και θεωρεί ότι τα έχει λύσει τα ζητήματα των γυναικών. Όχι, νομίζω ότι τα θέματα των γυναικών είναι σε καλά χέρια με τη Φιλανδική Προεδρία. Τρία θέματα που για την ομάδα μας είναι πολύ σημαντικά και Είχα και μία ερώτηση ε, για να ακούσω τη θέληση σας στη συνέχεια. Πρώτα απ' όλα, μιλήσατε για τη στρατηγική. Χρειάζεται στρατηγική για την ισότητα των φίλων στην Ευρώπη. Δεν χρειαζόμαστε μόνο κάποια έγγραφα εργασία, αλλά μια πραγματική στρατηγική για να δούμε πραγματικά τι πρέπει να ε, εφαρμοστεί στην πράξη και θα πρέπει να γνωρίζουμε και ξεκάθαρα τι θα γίνει με αυτά τα κράτη τα οποία δεν θα εφαρμόσουν ε, τα συμπεφωνημένα. Δηλαδή ε, δεν ε, θα πρέπει να μιλούμε για τις κυρώσεις μόνο αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα π.χ. με τα νητρόδη ή τα φωσφορικά στο έδαφος αλλά και για τα θέματα του γυναικών. Δεύτερο, Μιλήσετε για τη βία σε βάρος των γυναικών και μιλήσετε και για την προστασία των θυμάτων. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Είναι πολύ σημαντική η προστασία των θυμάτων, αλλά θύματα είναι όλες οι γυναίκες που έχουν πίσω τους ε, ένα τέτοιο συμβάν. Υπάρχουν όμως και ε, όλες εμείς οι γυναίκες που μπορεί να μην είμαστε θύμα κατά το παρελθόν, αλλά είμαστε ένας ε, ενδεχόμενος στόχος και νιώθουμε την απειλή, ακόμη και αν δεν έχουμε υποστεί κάποιο τέτοιο, κάποια τέτοια επίθεση μέχρι τώρα. Ένα λοιπόν το να είναι κανείς θύμα, αλλά υπάρχει και η γενική αίσθηση που έχουν πολλές γυναίκες στην κοινωνία μας ότι μπορούν να είναι ε, ένας δυνητικός στόχος βίας. Και σε ό,τι αφορά τα σεξουαλικά αναπαραγωγικά δικαιώματα, πράγματι υπάρχει πίεση και υπάρχει κάποια προσπάθεια να υπαναχωρήσουμε, να κάνουμε βήματα προς τα πίσω σε αυτά τα κεκτημένα μας ε, στον τομέα αυτό. Ελπίζω εσείς να υπερασπιστείτε τα σεξουαλικά αναπαραγωγικά δικαιώματα και να μην γίνει ούτε ένα βήμα προς τα πίσω όσο, όσο εσείς έχετε την Προεδρία. Πρόεδρε, σε ευχαριστώ πολύ. Σε μοίρα Ραφαέλα τώρα, Κύριε Ναχλητάν από την ομάδα των και Δημοκρατών. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ και για την ε, εισήγησή σας. Είμαι πολύ ευτυχής που η ισότητα των φύλων ε, εδώ θεωρείται προτεραιότητα είναι πολύ θετικό αυτό. Όμως ε, για τι γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια, γιατί το αναφέρατε αυτό και ε, χάρηκα που το κάνατε. όπω όμως είπατε, έχει κολλήσει το πράγμα και είναι σημαντικό να προχωρήσουμε. Θα ήθελα να γνωρίζω τι μπορείτε εσείς να κάνετε για να απεμπλακεί η κατάσταση. Ποιες είναι οι ενέργειες τις οποίες μπορείτε να προβείτε, γιατί είναι πολύ σημαντικό όντω να προχωρήσουμε και επίσης χρειάζεται να ε, δώσουμε εμείς το παράδειγμα στην Ευρώπη έχοντας ε, την ισότητα των φύλων στις υψηλότερες θέσεις και στις κυβερνήσεις ήδη πρόσφατα εμείς στην κάτω χώρες βρήκαμε μια λύση ε, και βασικά οι ενώσεις εργοδοτών και εργαζομένων και τα συνδικάτα ε, πρότεινε στην κυβέρνηση να, βάλουν, να βάλει στόχους ε, για την ισότητα, την ίση συμμετοχή ανδρών και γυναικών στις ανώτατες θέσεις και βλέπουμε ότι κάπως κινούνται τα πράγματα ήδη. Οπότε παρακαλώ να μου πείτε τι θα κάνετε εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Η και και Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ, ε, για την εισήγησή σας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εξωτερική πολιτική και αυτό που συμβαίνει σε άλλα κράτη-μέλη πολύ συχνά βλέπουμε να περιλαμβάνεται στα προγράμματα των κυβερνήσεών μας. Ε, δεν ενεργούμε, θέλω να πω, με τον ίδιο τρόπο σε εθνικό επίπεδο όπως σε ευρωπαϊκό. Χάρη όμως στις ΜΚΟ και στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών τα τελευταία χρόνια ακούμε όλο ένα και περισσότερο για βία, για απειλές κατά των γυναικών. Ε, κατά των γυναικών που προσπαθούν να υπερασπιστούν τις ελευθερίες τους. Οι γυναίκες αυτές οι οποίες υπερασπίζονται τα γυναικεία δικαιώματα ε, ε, δέχονται απειλές. Θα ήθελα να γνωρίζω λοιπόν πώς εσείς κύριε Πλόγκφιστ και η Φιλανδική Προεδρία θα χρησιμοποιήσετε την φωνή σας ε, στο ευρωπαϊκό και διεθνές προσκήνιο, ώστε να υπερασπιστείτε τις ευρωπαϊκές αξίες παντού ε, στην Ευρώπη αλλά και εκτός αυτής και για να υπερασπιστείτε τους ε, υπεραμεινόμενους των γυναικείων δικαιωμάτων εντός και εκτός Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Άντερσον. Εκτός μικροφώνου. ναι, Σα ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή σα παρέμβαση, κύριε Υπουργέ, που ήταν ενδιαφέρουσα σε μεγάλο βαθμό ε, και ίσως νομίζω στο σωστό δρόμο μπορούμε να συμφωνήσουμε. Ε, δύο-τρεις ερωτήσεις μου έρχονται τώρα στο μυαλό. Ουσιαστικά περί λεπτομεριών πρόκειται σε ό,τι αφορά τις γυναίκες στα δυτικά συμβούλια. Είπατε ότι θέλετε να το προχωρήσετε το θέμα και έχει δηλώσει και η κυρία Φοντρελόγεν την υποστήριξή σε αυτό το θέμα. Ερώτημα, τι μέτρα είστε έτοιμοι να ε, λάβετε ώστε πραγματικά να ισχύσει αυτή η εκπροσώπηση στα διοικητικά συμβούλια σε διάφορους τομείς ε, δεν υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση των γυναικών. Τι θα γίνει για τους τομείς αυτούς. Επίσης, ό,τι αφορά ε, την ε, ισότητα στην οικιακή εργασία κτλ. Τι συγκεκριμένα μέτρα προβλέπετε. Θα μπορούσατε να μας δώσετε κάποια παραδείγματα. Και κάτι άλλο που θα με ενδιέφερε είναι πώς θέλετε να εφαρμόσετε ή να ελέγξετε πράγματα τα οποία ουσιαστικά εκτελήσονται στο εσωτερικό οικογενειακό περιβάλλον. Και κάτι που είπε και η κυρία Νόιχελ, σωστά λέτε ότι θα πρέπει να μην παναχωρήσουμε καθόλου σε ό,τι αφορά την ε, προστασία των γυναικών, να μην υπάρχουν θύματα. Ε, οι γυναίκες ε, βλέπουμε ότι είναι σε χειρότερη θέση από ό,τι στο παρελθόν Έχουμε μέτρα, παραδείγματο χάρη, δημόσια ασφάλεια, αλλά ουσιαστικά δεν βλέπουμε οι γυναίκε ε, ε, ε, να νιώθουν πιο ασφαλεί. Αντίθετα, να νιώθουν ότι είναι πιο μεγάλε οι απειλέ. Τι μέτρα θα μπορούσατε να πάρετε εσείς για να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Από το ECR, λοιπόν, δεν βλέπω κάποιον συντονιστή από την ΚΟΕ ούτε και από αυτήν την ομάδα βλέπω, η Ευχένεια μάλλον. Ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ για την παρέμβαση αυτή. Και εγώ θέλω να συγχαρώ πως οι στις σας, οι την Φλανδική Προεδρία ε, σε ό,τι αφορά τώρα την ΚΟΕ, αυτό το οποίο εμάς ε, μας ανησυχεί είναι τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα. Θεωρούμε ότι ουσιαστικά είναι ένα έδος θεσμικής βίας σε βάρος των γυναικών. Το είπε και η συντρόφισσα. Μας ανησυχούν πάρα πολύ ε, τα, τα άτομα, γυναίκες που υπερασπίζονται τα δικαιώματα των γυναικών και στους Δήμους ε, και στις περιβαλλοντικές ενώσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για γυναίκες οι οποίες αντιμετωπίζουν ε, την εκμετάλλευση και στο πλαίσιο επιχειρήσεων που είναι και ευρωπαϊκές σε μεγάλο αριθμό τους. Ό,τι αφορά τώρα την ανισότητα και στο συνταξιδοτικό, βλέπουμε ακόμη να υπάρχει ένα χάσμα. Βλέπουμε να μην είναι ισομερής επίσης ε, η κατανομή των οικιακών εργασιών, ε, της φροντίδας, ε, είτε ηλικιωμένων είτε παιδιών. Και κάτι άλλο το οποίο μας ανησυχεί είναι και το ζήτημα της εμπορίας ανθρώπων και της ε, ε, πορνείας, της νόμιμης. Τι ε, θέλετε να κάνετε εσείς. Υπάρχουν μέρη στα οποία είναι ρυθμισμένη η πορνεία και βλέπουμε από την άλλη μεγάλη αύξηση της εμπορίας ανθρώπων. Σώμα Ευχαριστώ πολύ. Κάρεν τώρα, Μέλχερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να μιλήσω σε σχέση με τα όσα είπαν ε, προηγούμενοι μιλητές. Δυστυχώς δεν ακούγεται καλά η... η... Μάλλον δεν προβλέπεται ε, η διερμηνία από τα δανέζικα συγκεκριμένη συνεδρίαση. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, έπρεπε να το είχα πει. Παρασύρθηκα από τα Σουηδικά και άρχισα και εγώ να μιλάω στα Δανέζικα. Συγγνώμη, έχετε δίκιο. Ε, το, η διαφορά στις συντάξεις, ε, πώς θα εξασφαλίσετε ότι θα αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα και ότι θα έχουμε αρκετά στοιχεία ε, στη διάθεσή μας για να προχωρήσουμε. Μιλήσατε για τη σύμβαση της ε, Κωνσταντινούπολης. Υπάρχουν κράτη-μέλη που δεν την έχουν ακόμα κυρώσει. Έξι εξ αυτών ευρωπαϊκά κράτη-μέλη. Σε αυτή τη σύμβαση το άρθρο 33 μιλάει για ψυχολογική βία και την αναφέρει ρητά. Ξέρουμε πως η σωματική βία συχνά είναι αυτή που ακολουθεί την ψυχολογική βία. Θα ήθελα να ξέρω τι δουλειά κάνετε, συγγνώμη και πάλι από τους διερμηνήσεις και από όσους δεν καταλαβαίνουν τα δανέζικα. Ευχαριστώ. Δεν έχω κάποιον άλλον ε, στον κατάλογο των μητών. Α, ε, με το που το λέω βλέπω σηκώνονται κάποιες κάρτες. Ναι, παρακαλώ, εσείς έχετε το, λόγο. Merci. Monsieur le Ναι, σας ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Στη Γαλλία η επικαιρότητα ε, κινείται γύρω από την ε, γυναικοκτονία. Από την 1η Ιανουαρίου 109 γυναίκες έχουν ε, σκοτωθεί από τον σύντροφό τους ή από τον πρώην τους. Είναι ένας μεγάλος αριθμός και έχει διοργανωθεί μια ομάδα κρούσης για να βρεθούν λύσεις. Όπως ε, ξέρετε, υπάρχουν χώρες όπως και η Ελλάδα που εγώ έχω γεννηθεί, όπου δεν υπάρχουν καν στοιχεία. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω για αυτό το φαινόμενο ε, εσείς ε, τι σκοπεύετε να κάνετε στη διάρκεια της Προεδρίας σας. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Τώρα έκλεισε ο κατάλληλος των οπότε παρακαλώ κύριε Υπουργέ έχετε εσείς το λόγο. Κύριε Μπλόμκβιστ. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat edustajat. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ για τα εξαιρετικά και ενδιαφέροντα σχόλιά σας και για τις ενδιαφέρουσες ερωτήσεις σας. Θα προσπαθήσω να απαντήσω. Οι ερωτήσεις Ακολουθούν ε, γραμμές προβληματισμού που και εμείς ε, συχνά, που και εμάς συχνά μας απασχολούν. Ήταν πολλές ερωτήσεις, προσπάθησα να τις καταγράψω για να απαντήσω ε, σε όσες περισσότερες μπορέσω. Καταρχάς, ισότητα των φύλων. Και η ένταξη αυτού του θέματος σε όλες τις πολιτικές. Είναι ένα θεμελιώδης δικαίωμα και πρόκειται για μια αξία αλλά και για προϋπόθεση για ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή. Πιστεύουμε πως είναι σημαντικό να συνεχίσουμε την εργασία μας ώστε να προωθήσουμε μία διτή στρατηγική. Χρειάζεται στρατηγική για την ισότητα των φύλων στην Ένωση ε, που θα αποτελείται από μέτρα και από τη γενική προοπτική της ένταξης του διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές είναι σημαντικό να μπει το θέμα της ισότητας των φύλων στις οικονομικές πολιτικές και στις πολιτικές απασχόλησης και είμαι υπέρ της εντατικής συνεργασίας ανάμεσα στο Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Κομισιόν διότι αν θέλουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας για την ε, ένταξη του φύλου σε όλες τις πολιτικές χρειάζεται να ληφθούν μέτρα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Ευρωκοινοβούλιο έχει όντως εργαστεί εντατικά για να προωθήσει το θέμα της ισότητας των φύλων και μέσα στο πλαίσιο της λήψης αποφάσεων στην Ένωση. Υπάρχει θέμα όσον αφορά, ερώτηση μάλλον όσον αφορά τη στρατηγική υπερη Πιστεύουμε πως η στρατηγική της Κομισιόν, η οποία να είναι ισχυρή και πολύ σημαντική για τα επόμενα πέντε χρόνια, θα πρέπει να σχεδιαστεί αλλά και να αναλυφθεί πολιτική δέσμευση για την εφαρμογή των στόχων ισότητας Η στρατηγική αυτή είναι στην ατζέντα της Μελλοντικής Επιτροπής. Πρέπει να συνεχίσουμε αυτή τη διτή στρατηγική, ώστε να προωθήσουμε την ένταξη του θέματος της ισότητας των φύλων σε όλη την πολιτική. Η στρατηγική αυτή θα αποτελέσει μια καλή βάση για να αναπτυχθούν οι μελλοντικές μας πολιτικές ε, για την ισότητα των φύλων. Στη διάρκεια της Φιλανδικής Προεδρίας, συζητάμε την μελλοντική πολιτική περιισότητας μέσα στο Συμβούλιο Ισότητας, Απασχόλησης και Προστασίας του Καταναλωτή το Δεκέμβριο. Προβλέπεται η συζήτηση αυτού του θέματος για το Δεκέμβριο. Έγινε επίσης λόγος για τη βία και την ε, σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Σύντομα να πω γιατί πρόκειται για ένα εκτεταμένο πρόβλημα και θα μπορούσα επ' αυτού να μιλήσω το υπόλοιπο του χρόνου που μου αναλογεί. Η βία κατά των γυναικών είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα στην Ένωση και αυτό αφορά και τη χώρα μου, τη Φιλανδία. Πρόκειται για παράβαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, πρέπει να συνεργαστούμε ε, και να τηρήσουμε τις διεθνείς συμβάσεις μεταξύ αυτών και αυτήν της ε, Κωνσταντινούπολης ώστε να προλάβουμε και να δουλέψουμε κατά της βίας ενάντια στις γυναίκες εντός της ε, οικογένειας, της ενδοοικογενειακής βίας δηλαδή. Εμείς θέλουμε να καταπολεμήσουμε την βία χρησιμοποιώντας ε, τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και όπως είπα ήδη η Φιλανδία στηρίζει εντόνως τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης στη διάρκεια της ε, προεδρίας μας ε, δε θα θέλαμε να ενθαρρύνουμε όλες τις χώρες που δεν έχουν κυρώσει την σύμβαση αυτή να προβούν στην κύρωσή της. Επιπλέον θα θέλαμε να προωθήσουμε ε, την κύρωση της συνθήκης της ε, Κωνσταντινούπολης από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. όσον αφορά την πρόθεση των δικαιωμάτων των θυμάτων ε, βίων εγκλημάτων και αυτό είναι πολύ θυματικό θέμα, θα υπάρξουν συμπεράσματα του Συμβουλίου για τα δικαιώματα των θυμάτων στη διάρκεια της Προεδρίας μας. Προσπαθώ, όπως είπα, να απαντήσω σε όσο γίνεται περισσότερες ερωτήσεις, γι' αυτό και οι απαντήσει μου είναι σχετικά σύντομες. Υπήρξε και μια ερώτηση για τις γυναίκες και μάλλον για τα δικαιώματα ε, των γυναικών και των κοριτσιών, καθώς και ε, τα αναπαραγωγικά και σεξουαλικά δικαιώματα. Στη διάρκεια της ε, Φιλανδικής Προεδρίας θεωρούμε πως αυτά τα δικαιώματα είναι οριζόντιες προτεραιότητες. Θέλουμε να χειραφετήθουν οι γυναίκες, να προωθήσουμε κοινωνικές προδιαγραφές, να δουλέψουμε πάνω στα κοινωνικά στερεότυπα, να ε, επανέλθουμε στο θέμα της σεξουαλικής παρενόχλησης αλλά και να ε, τονίσουμε τις ανάγκες των γυναικών και κοριτσιών με ε, ειδικές ανάγκες. Υπάρχει και το θέμα μιας πρότασης που αφορά τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια, η οποία έχει παγώσει από το 2011 Έχω, έχει συζητηθεί το, θέμα, στη διάρκεια αυτής της περίοδου και είναι πιθανό η μελλοντική πρόεδρος της Επιτροπής να θεωρήσει πολύ σημαντική την προώθηση αυτού του θέματος. Η Φιλανδία στη διάρκεια της Προεδρίας της θα προσπαθήσει και θα καταβάλει όλες τις απαραίτητες προσπάθειες. Ωστόσο, για να είμαι ειλικρινής, θα πρέπει να σας πω ότι δεν ε, απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία για αυτό το θέμα στο Συμβούλιο. Το κείμενο του, του, εισοδικίας είναι έτοιμο προς υιοθέτηση εάν διαπιστώσουμε πως υπάρχει δυνατότητα. Γι' αυτό ελπίζουμε πως θα το καταφέρουμε. Υπάρχει και το θέμα των μαχητών Τη ελευθερία, ε, δηλαδή των υπερασπιστών ε, των γυναικείων δικαιωμάτων. Ε, ο Υπουργό Εξωτερικών της Φιλανδίας διοργάνωσε συνέδριο σε σχέση με την κατάσταση των υπερασπιστών των γυναικείων δικαιωμάτων και πώς θα μπορούσαμε να τι προστατεύσουμε, καθώς πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και θα θέλαμε να συζητήσουμε και να προωθήσουμε το θέμα αυτό. υπήρξε και ένα θέμα σε σχέση με την ε, διακίνηση γυναικών και την πορνεία. Ε, ερώτηση δηλαδή. Πιστεύουμε πως είναι σημαντικό να θεωρηθεί η διακίνηση γυναικών ως μια μορφή βίας κατά των γυναικών. και να θεωρηθεί ως ε, ένδειξη διακρίσεων επί τη βάση του φύλου. Οι περισσότεροι που πέφτουν θύματα διακίνησης στην Ευρώπη τη σήμερα ημέρα είναι γυναίκες και κορίτσια. Στηρίζουμε λοιπόν ε, το συντονίστρια τη οποία η εργασία γίνεται πάνω στην οδηγία για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να συντονίσουμε και ε, την εργασία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού καθώς και την ε, δουλειά που γίνεται στα κράτη-μέλη για την εφαρμογή της οδηγίας. Βεβαίως είναι ανησυχητικό να διαβάζει κανείς την έκθεση της ε, Μίριαμ Βασιλιάδου που λέει ότι Οι μισές από τις γυναίκες που διακινούνται προορίζονται για σεξουαλική εκμετάλλευση και ότι τα δύο τρίτα της διακίνησης ανθρώπων είναι γυναίκες. Είναι ένα φαινόμενο όπου χαρακτηριστικά βλέπουμε να επηρεάζεται από το φύλλο. Το θέμα το ίσης αμοιβή είναι εξίσου σημαντικό και στην Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπουμε ότι διαονίζονται οι διαφορές ε, αμοιβών ε, μεταξύ ανδρών και γυναικών. Θα πρέπει λοιπόν και στα κρατημέλη να γίνει ε, επισταμένη προσπάθεια ώστε να εξισωθούν οι αμοιβέ αλλά και οι συντάξεις. Η Φιλανδία λοιπόν θα φέρει αυτούς τους στόχους ε, στο Συμβούλιο και θα προσπαθήσει να τους περιλάβει στη, στα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Αυτά λοιπόν, προσπάθησα να καλύψω όλες τις ερωτήσεις. Λυπούμε εάν δεν απάντησα σε όλους σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά κύριε Υπουργέ. Νομίζω ότι απαντήσατε πάρα πολύ, ε, με πολύ πλήρη τρόπο. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ε, εύχομαι, αλλά ταυτόχρονα εύχομαι και σε όλες και όλες μας ε, ε, καλή επιτυχία στην εφαρμογή των ε, προτάσεών σας και ελπίζω να τα ξαναπούμε στο διάρκεια του εξαμήνου. Καλή δουλειά. Τακ. <laughs> So, κυρίε uh, κυρίες και κύριοι, προχωρούμε στο επόμενο σημείο της ημερήσια διάταξης και συγκεκριμένα σε μια ακρόαση, μια ανταλλαγή απόψεων με πολύ γνωστά ευτυχώς πρόσωπα, την Edith Bauer και τον Μίκαλ Γκούσταυσον, το θέμα αυτής της ακρόασης είναι το Σώμα Εμπειρογνωμών για το ΕΓΚΕ, το Ινστιτούτο Ισότητας Φίλων, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο, θα ακούσουμε την παρουσίαση και μετά θα έχουμε τη δυνατότητα να θέσουμε τις ερωτήσεις μας. Και έχουμε τώρα σε αυτό το σώμα ε, συναδέλφους ε, οι οποίοι είναι πολύ πεπειραμένοι στα θέματα αυτά και επομένως μπορούν να εκπροσωπήσουν ε, καλά και το Κοινοβούλιο. Women first, men first. Εντάξει, κύριε Γκούσταυσον, πρώτα εσείς και μετά κυρία Μπάουρ. Καλώς ήρθατε και δύο. Hej Eh, Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα θέλαμε σύντομα να σας κάνουμε μια ενημέρωση. Καταρχάς ε, να σας πω περί τίνος πρόκειται, ποιος είναι αυτό ο φορέας, ποιο είναι αυτό το σώμα εμπειρογνωμόνων. Δεν θέλω να μακρηγορήσω βέβαια αλλά καλό θα ήταν ε, να ε, γίνει κατανοητό για τι είδους οργάνωση μιλάμε. Σε τι οργάνωση ανήκει η και εγώ. Εγώ, όπως γνωρίζετε, Είμαι ένας άνθρωπος ε, που αγαπά πολύ τη μητρική γλώσσα. Μιλάω πάρα πολύ καλά, ε, με πολύ μεγάλη χαρά τη δημητρική μου γλώσσα. βέβαια όταν έχω γράψει την παρουσίαση αυτή στα ε, αγγλικά και πρέπει να μιλήσω ειδικά δεν είναι και τόσο εύκολο οπότε θα μου επιτρέψετε ζητώντας και συγγνώμη από τη δική καμπίνα από εδώ και πέρα να συνεχίσω στα αγγλικά. συντομία λοιπόν, θα ήθελα να σας μιλήσω για το ΕΓΚΕ, που είναι ένα φόρουμ εμπειρογνωμόνων. Θα μιλήσω για την οργάνωση και θα σας πω και για το 2019 τι προβλέπουμε. Καταρχάς, μπορεί να το ξέρετε βέβαια, αλλά θα σας το επαναλάβω. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση 44 Οργανισμή, η ΕΙΓΚΕ είναι ένα από αυτού του οργανισμού, είναι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ισότητα των Φύλων. Όλε αυτέ ε, οι οργανώσει ανεξάρτητε και χρηματοδοτούνται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, παρέχουν δε πληροφορίες, συμβουλές για την ε, λήψη αποφάσεων και χάραξη πολιτικής και επίσης εκτελούν καθήκοντα από τους αναθέτω κατημέλη μέλη Τι κάνει το ΕΙΓΕ. Πρώτα απ' όλα, ιδρύθηκε το 1999. Στη Σουηδία τότε τονίστηκε ότι είναι ανάγκη να υπάρχει ένας τέτοιος οργανισμός για την ισότητα των φύλων. Χρειάστηκε βέβαια λίγος καιρός ε, μετά από αυτό, γιατί πρώτα έπρεπε να γίνει μια μελή της Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρότεινε το 2004 να ιδρυθεί πράγματι ένας τέτοιος οργανισμός και η απόφαση από την Κομισιόν ελήφθη το 2005. Το 2006 αποφασίστηκε ότι η έδρα του Ινστιτούτου θα είναι το Βίλνιους. Επίσης εγκρίθηκε τότε και ο κανονισμός του Κοινοβουλίου και του Συμβούλου και το 2007 ορίστηκε το πρώτο δικτικό συμβούλιο του Ινστιτούτου. ως φορέας λοιπόν της Ένωσης, το ΕΓΚΕ ουσιαστικά λογοδοτεί αφενός στο Διοικητικό του Συμβούλιο και αφετέρου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κάτι άλλο που ενδεχομένως το γνωρίζετε, έχω εργαστεί και εγώ πολλές, πολλά χρόνια ε, και γνωρίζω ότι η ισότητα μεταξύ των γυναικών είναι θεμελιώδης αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα στόχος μας είναι η ισότητα μεταξύ των ανδρών και των γυναικών να γίνει πραγματικότητα για όλους τους Ευρωπαίους αλλά και όχι μόνο. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο ε, Πληροφοριών για την ισότητα των δύο φύλων. Ποια είναι τώρα η δομή του έγκε? Τριμερής θα έλεγα. Δηλαδή φυσικά υπάρχει το Διοικητικό Συμβούλιο Υπάρχει ο διευθυντής, ε, το τελεστικό δηλαδή, εκτελεστική εξουσία και έχουμε και το σώμα των εμπειρογνωμόνων. Εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ, γιατί αποφασίστηκε εγώ και Edith Bauer να είμαστε τα δύο μέλη που θα εκπροσωπούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το σώμα εμπειρογνωμόνων είναι το συμβουλευτικό ε, σώμα του Ινστιτούτου. Δεν ξέρω αν μπορείτε να διαβάσετε τις διαφάνειε, γιατί είναι μικρά τα γράμματα. Ή εγώ γέρασα τέλος πάντων. Πάντως εγώ δεν τα πολύ διαβάζω. Ή και τα δύο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, η βασική ε, αρμοδιότητα του σώματος είναι παρέχει τεκμηριωμένη γνώση στον τομέα της ισότητας των φύλων να απαρτίζεται από ένα πλήρες και ένα αναπληρωτικό μέλος από κάθε κράτος μέλος, δύο μέλη ε, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τρία ε, μέλη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από διαφορετικέ οργανώσεις. Το Σώμα Επιρογνωμόνων στηρίζει το Διευθυντή για να εξασφαλιστεί αριστεία και ανεξαρτησία των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου και εξασφαλίζει τη στενή συνεργασία μεταξύ του Ινστιτούτου και των διαφόρων αρμοδίων φορέων και οργανισμών των κρατών μελών. Κανονικά έχουμε κάποιες σχέσεις με διάφορους ε, ενδιαφερομένους φορείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τον αρμόδιο επίτροπο και με τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΤΖΑΣΤ Με το Συμβούλιο έχουμε επαφή με τις Προεδρίες και τα κρατημέλη και σε ό,τι αφορά το Κοινοβούλιο έχουμε επαφή με την Επιτροπή Γυναικών και άλλες ε, επιτροπές ε, ε, αρμόδιες για τα εκάστοτε ζητήματα που μας απασχολούν. Ποια είναι η δομή του ΕΙΓΕ. Τώρα είναι ακόμα πιο δύσκολο να διακρίνεται. Ούτε στο iPad δεν ξέρω αν τα βλέπω καλά εγώ. Λοιπόν, έχουμε το διευθυντή που είναι επικεφαλής ε, του Ινστιτούτου και έπειτα έχουμε τρία τμήματα, τη διοίκηση, τις επιχειρήσεις και τη διαχείριση γνώσεων και επικοινωνία. Και υπάρχουν και μονάδες που υπάγονται ε, στο δεύτερο με επιχειρήσεις, operations και στο άλλο, στο τρίτο τμήμα. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, έχουμε όμως το πρόγραμμα εργασίας μας για τη φετινή χρονιά το 2019, το οποίο εστιάζει σε τέσσερα σημαντικά ζητήματα. Είναι η, ένταξη, η ενσωμάτωση της διάστασης του φίλου σε όλες Ένα, δύο είναι στατιστικές δείκτες. Το τρίτο είναι η βία λόγω φύλου και το τέταρτο είναι η διαχείριση γνώσεων και επικοινωνία. Περισσότερες πληροφορίες φυσικά μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο, στο facebook ε, ή οπουδήποτε. Μπορείτε λοιπόν να έρθετε σε επαφή μαζί μας. Αυτό είναι το υπόβαθρο. Για να καταλάβετε για ποιο λόγο εμείς είμαστε εδώ. Είμαστε υπόλογοι σε εσά. Εσά ε, εκπροσωπούμε, μα επιλέξαν να σα εκπροσωπούμε στο Σώμα Εμπειρογνωμών, άρα λογοδοτούμε σε εσά. Edit, μπορείς να συνεχίσει. Ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι και πάλι εδώ μαζί σας ε, σήμερα. Ήμουν μέλος ε, της Επιτροπής για 10 χρόνια και είμαι περήφανη που ακούω τον Υπουργό να συζητά για την οδηγία για τη διακίνηση ανθρώπων, διότι ήμουν εισηγήτρια για αυτή την οδηγία ε, και ήμουν εισηγήτρια για πολύ και διαφορετικά θέματα και άρθρα, αλλά χαίρομαι γιατί αυτή ήταν μία ε, έκθεση η οποία έγινε πριν ε, ε, να υπάρξει νομοθεσία για το μισθοδοτικό χάσμα ανδρών και γυναικών. Χαίρομαι επίσης και είμαι περήφανη που εξελέγει ε, μέλος ε, του Φόρου Εμπεριγνωμένων. Ήταν πραγματικά ε, μια πάρα πολύ καλή περίοδος και είναι το, το λίκνο αυτού του θεσμικού οργάνου και θυμάμαι πόσο δύσκολα ξεκίνησε αυτό το Ίδρυμα. σκεφτείτε ότι για δύο χρόνια υπήρχε μόνο ένας διευθυντής και ένας γραμματέας και τίποτα άλλο. Περιμέναμε λοιπόν πέντε χρόνια περίπου για να μπορέσουμε να το δημιουργήσουμε αυτό το Ίδρυμα και νομίζω ότι μπορώ να πω με ικανοποίηση ότι το Ίδρυμα αυτό οδηγεί σε πολύ καλά αποτελέσματα results and, and uh, achievements και εξαιρετικά επιτεύγματα. I will Και επειδή υπάρχει και διερμηνία, από εδώ και πέρα θα συνεχίσω στα σλοβακικά. Για να πω κάποιες περισσότερες πληροφορίες ε, για το Φόρουμ των Εμπειρογνωμόνων, κυρίως ε, για τα όσα κάνει η ομάδα εργασίας για τα θέματα ισότητας του φύλου και το σχετικό δίκτυ. Ο δίκτυς ισότητας φύλου Αυτός ο δείκτης είναι ίσως ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα που έχουμε ε, καταφέρει σε αυτό το Ινστιτούτο. Φανταστείτε ότι πρέπει να ε, συμπηλήσετε όλους αυτούς τους δείκτες. Ε, έχουμε 31 διαφορετικούς δείκτες που ουσιαστικά αφορούν έξι θεματικούς τομείς, την απασχόληση, τα οικονομικά της γνώσης, το χρόνο, τη δύναμη, την ισχύ, ε, που δεν μ' αρέσει και πολύ σαν λέξη τέλος πάντων, ε, ίσως πολιτική ισχύ θα ήταν καλύτερη, πολιτική εξουσία και υγεία. Αυτή είναι η εξταματική τομή. Και έχουμε κάποια δορυφορικά θέματα, όπως είναι η βία σε βάρος των ε, γυναικών και οι ανισότητες ποιο είναι το βασικό καθήκον ε, και πόσο δύσκολο είναι το εγχείρημα. Αν δει κανείς τις στατιστικές που υπάρχουν σήμερα, διαπιστώνεται εύκολα ε, τι δυσκολίες υπάρχουν. Έχουμε το μισθολογικό χάσμα, ε, όμως ε, τα στοιχεία είναι από δύο χρόνια πριν ε, και ε, υπάρχει αντίθεση σε σχέση με το τι γίνεται ε, στην Ένωση. Δηλαδή παίρνετε απαρχιωμένα στοιχεία πολλές φορές ή στοιχεία τα οποία δεν έρχονται από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία. Soft data όπως τα λέμε. Πρόκειται για στοιχεία τα οποία προέρχονται από διάφορες ε, δημοσκοπήσεις ε, και καταλήγουν ε, τα απορίσματα σε κάποιους δείκτες. Ας πούμε, το στο του Δουβλίνου, το έδραμα του Δουβλίνου μας δίνει κάποια πληροφορία. Εσύ, το ΦΡΑ, ο οργανισμός δηλαδή ε, και Και Έχουμε κάποια στοιχεία σε ό,τι αφορά τη βία ε, σε βάρος των γυναικών. Τα στοιχεία που έχουμε το 2012 και δεν ξέρουμε πότε θα έχουμε πιο επικαιροποιημένα στοιχεία, άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να επικαιροποιήσουμε τα στοιχεία που έχουμε του θεματικούς αυτούς τομείς. Επομένως, αυτό το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας και αυτό το οποίο κάνουν οι υπάλληλοι ε, στην ε, υπηρεσία μας είναι ουσιαστικά κάτι που θα έλεγα προσεγγίσει στο θαύμα. Υπάρχουν πολλά προβλήματα που άπτονται της ε, κατάρτισης δικτών και της συγκέντρωσης των αποτελεσμάτων. Υπάρχουν επίσης διάφορες ε, ε, ομάδες εργασίας, αυτό το σώμα εμπειρογνωμόνων που προσπαθεί να λύσει αυτά τα προβλήματα. Τρία χρόνια έχω εργαστεί ομάδα εργασία, ε, διατέλεσα και πρόεδρος, επανεξελέγει τώρα και είναι και μέλος και ο Μίκαλ Γκούσταυσον. Στο τέλος τώρα να πω κάτι ακόμη αν μου επιτρέπετε πάρα πολύ σημαντικό πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό είναι να καταρτιστούν αυτοί οι συνθετικοί δείκτες. Ε, γιατί πολλές φορές μιλάμε για ισότητα, αλλά αοριστολογούμε. Όταν όμως κάνουμε σύγκριση και καταρτίζουμε δείκτες, τα πράγματα αποκτούν ε, μια πιο σαφή εικόνα. αν μιλάμε 66,2 στα 100 ή κάτι τέτοιο, μιλάμε πιο πολύ για κάποιες τάσεις, αλλά δεν μπορούμε να αυταπατώμεθα ότι μόνο προς τα εμπρός πηγαίνουμε και βελτιώνουμε την κατάσταση από χρόνο σε χρόνο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Για παράδειγμα, από το 2005 για το θεματικό τομέα χρόνος έχουν ε, ε, επιδεινωθεί οι στατιστικές. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Έχουμε διακοιμάσει από το 50 έως το 82. 50 είναι Ελλάδα, 82 είναι η Σουηδία για παράδειγμα σε ό,τι αφορά αυτούς τους δείκτες. Θα ήθελα τώρα να σας πω και κάτι άλλο. Τα τρία τελευταία χρόνια έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις και διάλογο. Ένα πολύ σημαντικό θέμα που μας απασχόλησε είναι η βία σε βάρος των γυναικών, κάτι το οποίο ακούσαμε και προηγουμένως. Έχουμε στοιχεία, έχουμε ένα δείκτη για τις 27 Εμείς δεν θέλουμε να έχουμε, ε, παραδείγματο χάρη, άνοδο του στοιχείου για του άντρε. δηλαδή να έχουμε βία σε βάρο αντρών, είτε έχουμε αυτό το 27 και δεν σημαίνει ότι θα θέλαμε να αυξηθεί για του άντρε. Εμείς θέλουμε να μην υπάρχει βία σε βάρο κανενός από τα δύο φύλλα. «90 προς 5 είναι η αναλογία. Όλα αυτά τα στοιχεία ενσωματώνονται, υποτίθεται, στο βασικό δίκτυο. Γιατί δεν γίνεται αυτό όμως. Πρώτον δεν έχουμε γραμμικά στοιχεία ε, για να επεξεργαστούμε. θα πρέπει να είχαμε χρονοσυρές, ε, αλλά δεν έχουμε, γιατί από το 2012 και μετά δεν έχουμε νέα στοιχεία, όπως σας είπα. Επίσης ένα σημαντικό ζήτημα είναι και η αξιοπιστία αυτών των δεδομένων. Για να έχουμε πραγματικά αξιόπιστους δείκτες πρέπει να είναι αξιόπιστα και τα στατιστικά στοιχεία. Δεν το έχουμε πάντα αυτό όμως. Δηλαδή πολλές φορές ε, δεν ανταποκρίνεται το στοιχείο ε, που έχουμε, το νούμερο που έχουμε με αυτό το οποίο μετρήθηκε στην πράξη, ό,τι αφορά την ε, βία για παράδειγμα. Υπάρχουν πίσω και πολλά άλλα πράγματα. Μπορεί να θεωρούμε ότι έχει να κάνει με άσκηση βίας, αλλά τελικά μετράμε κάτι τελείως διαφορετικό π.χ. την ε, πιστοσύνη στο δικαστικό σύστημα, την πιστοσύνη στην αστυνομία. Και αυτοί είναι δείκτες. που δημιουργούν μεγάλες ε, διαφοροποιήσεις στο τελικό αποτέλεσμα. Άρα, σε ό,τι αφορά τη βία, ε, Μπορεί να φαίνεται π.χ. ότι στη Σουηδία είναι πολύ τη βία σε σχέση με τις χώρες των Βαλκανίων ή το ανάποδο. Υπάρχουν μεγάλες διαφοροποίησεις. Γιατί, επαναλαμβάνω, πολλές φορές μετράμε τελείως διαφορετικά πράγματα από χώρα σε χώρα με αυτά τα στοιχεία, άρα δεν μπορεί να υπάρξει συγκρισιμότητα δεν έχουμε καταφέρει να βρούμε έναν διορθωτικό συντελεστή, να διορθώσουμε ενδεχομένως κάποιες ανακρίβειες ώστε να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα οι δείκτες αυτοί, τα στατιστικά αυτοί, Και αυτό ήταν και το βασικό στοιχείο που μας είχε απασχολήσει, σε ό,τι αφορά δηλαδή την ενσωμάτωση των στατιστικών ε, στους βασικούς δείκτες. Ε, δεν μπορεί να γίνει αυτό δυστυχώ. Γι' αυτό και έχουμε προχωρήσει σε μια διαφορετική μεθοδολογία. Intersect inequalities λέγεται στα αγγλικά, αυτό το οποίο θέλω τώρα να σχολιάσω. Είναι ένα άλλο πρόβλημα με το οποίο έχουμε να κάνουμε. Όταν μιλάμε, παραδείγματο χάρη, για τον τόπο γέννηση, ε, έχουμε να λάβουμε υπόψη και άλλα στοιχεία. Το μεταναστευτικό, για παράδειγμα. Ε, δεν μας ενδιαφέρει που γεννήθηκε κάποιος ε, στη Βουδαπέστη ή στο Άμστερνταμ, για παράδειγμα. Αλλά τι γίνεται με αυτούς που γεννήθηκαν στην Ένωση ή αυτούς που έχουν γεννηθεί σε μια τρίτη χώρα. πάντα στόχος είναι η ενσωμάτωση των στοιχείων, όπως είπα, στο βασικό δίκτυ. Δυστυχώς πάλι τα αποτελέσματα εδώ δεν ε, είναι απόλυτα αξιόπιστα. Έχουμε να κάνουμε πολλά προβλήματα και αυτά μας απασχολούν και σε ομάδες εργασίας. Παραδείγματος χάρη έχουμε προβλήματα πολιτικά, προβλήματα μεθοδολογικά αλλά πρόκειται για ένα πολύ ενδιαφέρον για εμάς ζήτημα και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούν να χρησιμοποιούνται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά τα στοιχεία. Μέχρι πρόσφατα η Κομισιόν χρησιμοποιούσε στοιχεία τα οποία παίρναμε από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά την δουλειά που κάνουμε στο Ινστιτούτο και στο Σώμα Εμπειρογνωμόνων και πραγματικά νομίζω ότι πρέπει να αναβαθμιστεί ε, η εικόνα για την ε, δουλειά που κάνουμε και να έχετε πλήρη αίσθηση του πόσο δύσκολο είναι το έργο μας. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γκούρστασον έχει κρεματίσει και πρόεδρο τη μας κατά το Λοιπόν, να δώσω τώρα το λόγο στου συναδέλφου. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση, κυρία Μέλχιο. Το βρίσκω λίγο ανησυχητικό το γεγονός ότι υπάρχουν τέτοια προβλήματα για τα δεδομένα για το δίκτυο. Πώς μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι έχουμε τα στοιχεία που χρειαζόμαστε για τον δίκτυο που επιθυμούμε. Για παράδειγμα, τα στοιχεία για τη βία κατά των γυναικών είναι 7 ετών, από το 2012. Και θα ήθελα να μου πείτε και λίγα περισσότερα πράγματα για το πώς μπορούμε να εξορθολογήσουμε και το έργο του οργανισμού. Διότι φαίνεται να είναι ξεχωριστή από τις άλλες ε, υπηρεσίες και οργανισμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να έχουμε περισσότερα από όσα κάνει ο οργανισμός, ώστε να ε, παίρνουμε και περισσότερα για τα χρήματα που ε, δαπανούμε για τον οργανισμό αυτό, αλλά αυτό σημαίνει και εξορθολογισμό των εργασιών. Ευχαριστώ η Σαμίρα Ραφαέλα. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Δύο ερωτήσεις. Η μία είναι οι διάφορες ε, ε, ενότητες. Χαίρομαι που το αναφέρατε, αλλά θα ήθελα να ξέρω πώς θα ε, εξασφαλίσετε ότι έχετε αρκετά εύρος δεδομένων και αρκετή, αρκετά ποιοτικά δεδομένα, ώστε να στοχεύσετε συγκεκριμένα θέματα τα οποία αφορούν διάφορες γυναίκες. Διότι όταν συζητούμε για τις γυναίκες, ναι, συζητούμε για τις γυναίκες, αλλά υπάρχουν πολλές και διαφορετικέ γυναίκε. Είμαστε διαφορετικέ μεταξύ μα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε δεδομένα ώστε να υπάρχει συγκεκριμένη καλή προσέγγιση για γυναίκε με τελείω διαφορετικό υπόβαθρο. Ε, εδώ έχουμε επίσης και το θέμα της βίας ε, ε, λόγω φύλου. Έχουμε για παράδειγμα στο διαδίκτυο παρενόχληση, εκφοβισμό γυναικών, ακόμα και βία λοιπόν ε, μπορεί να έχουμε στα επόμενα χρόνια και είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να εστιάσουμε στη συνέχεια. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν τι μπορείτε να κάνετε εσείς για το θέμα αυτό από την πλευρά της έρευνας και της ε, μελέτης των θεμάτων αυτών. Ευχαριστώ. Μόνικα Βάνα. Ευχαριστώ κυρία. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι που σας βλέπω κυρία Γκούσταυσον και κυρία Μπάουερ. Εμείς ως πράσινε ε, υποστηρίξαμε πολύ το έργο του ΕΙΓΕ τα τελευταία χρόνια, διότι εμείς ως ευρωβουλευτές βασιζόμαστε σε καλέ δεδομένα ε, και προσβλέπουμε στην καλή συνεργασία και το επόμενο διάστημα σε αυτή τη φοιτεία. Έχω και μία ερώτηση γιατί είμαι και στην Επιτροπή Προπολογισμών και στην Επιτροπή Περιφερειακή Ανάπτυξη. Ιδιαίτερα στην Περιφερειακή Ανάπτυξη, όταν συζητούμε περιφερειακά κονδύλια και ε, περιφερειακέ πολιτικέ, δεν έχουμε στοιχεία για την ισότητα των φύλων αναπεριφέρεια και είμαι αρμόδια για την ε, ε, πολιτική συνοχή και θέλουμε να έχουμε μια τροπολογία, να έχουμε δηλαδή δεδομένα για το φύλλο, διότι υπάρχει μεγάλο μερίδιο του προπολογισμού που δίνεται στα θέματα αυτά. Θα μπορούσατε να μας πείτε λοιπόν τι κάνετε εσείς με περιφερειακά δεδομένα και αν θα μπορέσουμε να έχουμε ε, πρόοδο τελικά στην περιφερειακή πολιτική. Ευχαριστώ η Έλλης και μετά η Λίνα. Νομίζω ότι είχα δώσει το χρόνο μου στη συνάδελφο, αλλά θα ήθελα να σχολιάσω κι εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις παρουσιάσεις και εγώ θα ήθελα να ρωτήσω πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε ότι τα δεδομένα τα οποία χρησιμοποιείτε είναι αντίστοιχα με τα δεδομένα των κρατών μελών, ώστε να μην κάνουμε τα ίδια πράγματα. Εγώ ως πρώην Υπουργός διαπίστωσα ότι δυστυχώς πολύ συχνά και αρκετά καθυστερημένα υπάρχει κάτι το οποίο διερευνούσαμε ε, και εγώ θα ρωτούσα στον οργανισμό και ήταν αρμοδιότητα του δικού μου Υπουργείου, συνέβαινε σε άλλη χώρα και υπήρχαν στοιχεία και επομένως θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε στο παρελθόν ή κάπως να μάθουμε και για κάποια πράγματα. Τι κενά λοιπόν υπάρχουν και τι θεωρείτε ότι θα μπορούσαν να κάνουν οι χώρε μελή καλύτερα, ώστε τα στοιχεία τα οποία παράγετε εσεί ε, να μπορούν να χρησιμοποιούνται στη χάραξη πολιτική και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στι χώρε μέλη. Ευχαριστώ πολύ. Η Λίνα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ρωτήσω κι εγώ κάποια πράγματα αντίστοιχα με τα θέματα που μόλις ακούστηκαν and Eurostat as well, because I think... Νομίζω ότι βασίζεστε και στα στοιχεία της Eurostat, αν δεν κάνω λάθος. Διότι ό,τι κάνετε όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία για το φύλλο είναι κυρίως ε, ε, διαχωρισμός των στοιχείων μεταξύ των φύλων. Αλλά ε, είναι κυρίως ανδροκεντρικά τα στοιχεία αυτά και θα ήθελα να ξέρω λοιπόν τι κάνετε προκειμένου να εξασφαλίσετε ότι γίνεται διαχωρισμός μεταξύ των δύο φύλων Υπάρχει και το θέμα της χρονικής συγκυρίας των στοιχείων και κάποια από τα βασικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας προκειμένου, για παράδειγμα, να ε, μετρήσουμε την αμυστή εργασία και να μετρήσουμε την ανισότητα μεταξύ των φύλων σε τέτοιες περιπτώσεις εργασίας αμυστή, δεν έχουμε στοιχεία ε, για κάθε χώρα ε, στην ίδια χρονική συγκυρία. Δεν έχουμε δηλαδή κάποια χρονική ακολουθία να ακολουθήσουμε. Ε, θα ήθελα να ξέρω λοιπόν τι κάνετε με τη Eurostat και θα ήθελα να ε, πιέσουμε και τη Eurostat να ε, συμμετέχει σε διεθνή φόρουμ ε, για στατιστικά στοιχεία. Για παράδειγμα, στα Ηνωμένα Έθνη διοργανώνουν σε διάφορα μέρη του κόσμου την τελευταία 15 είχαν τουλάχιστον 7 παγκόσμια φόρουμ για ε, στατιστικά στοιχεία για το φύλλο και από ό,τι ξέρω η Eurostat δεν ήταν παρούσα σε καμία από αυτές τις συνεδριάσεις. Βλέπετε λοιπόν ότι θα πρέπει να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε κάπως αυτό το ανδροκεντρικό στατιστικό σύστημα. Θα πρέπει λοιπόν να πιέσουμε πάρα πολύ την Eurostat εάν πραγματικά επιθυμούμε να βρούμε μια λύση για τα προβλήματα ε, τα οποία μας ε, περιγράψατε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Η Ρώσα Φεραγκούτ και μετά η Μαριανόχη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Και Έρικα, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Καλή φίλη από τότε που ήσουν ε, εδώ και είχες μια πολύ σπουδαία ε, θέση και μεγάλη επιτυχία. Από ό,τι φαίνεται έχει γίνει μια μελέτη για τη γυναίκα στον ψηφιακό κόσμο. Μπορείτε να μας πείτε κάτι για αυτή τη μελέτη και να όχι να μας την φέρετε εδώ, γιατί εκεί φαίνεται πως υπάρχουν στοιχεία για τις τάσεις στον ψηφικό κόσμο σε θέματα φύλου ότι υπάρχουν ε, τάσεις όπως το body shaming ή το sexting και διάφορα άλλα που μπορεί να αποτελούν ε, βία. Επίσης να δούμε τι γίνεται με την απασχόληση, ε, τι γίνεται με την παιδεία, με τα θέματα φύλου και αναπηρίες. Η Μαρία Ευχαριστώ πολύ για τις παρουσιάσεις και όταν ε, μιλάμε και για τον ε, προπολογισμό πάντα τονίζουμε και το θέμα ε, αυτό είναι πολύ σημαντικό και η δουλειά σας. Δεν έχουμε καταφέρει 5-10 χρόνια τώρα να έχουμε καλά στατιστικά στοιχεία και επιστημονικά τεκμηριωμένα που τα χρειαζόμαστε όμως γιατί πρέπει να μπορούμε να καταρρύπτουμε και να διαψεύδουμε και τις ψευδείς ειδήσει. Γι' αυτό ακόμη πιο χρήσιμα είναι αυτά τα αξιόπιστα δεδομένα. Συγκεκριμένα λοιπόν, ε, τι κάνετε με τις ψευδείς ειδήσει που διαδίδονται στην Ευρώπη. Παραδείγματος χάρη, ε, μόνο από το τότε που υπάρχουν πρόσφυγες, ε, είναι μια πολύ ξεκάθαρη ψευδισίδηση, έχουμε βία σε βάρος των γυναικών. Αυτό είναι μια ανοησία. Ε, ούτε αυτή τα εγκλήματα τιμής, για παράδειγμα, ε, δεν γίνεται μόνο με όσους έχουν με λαψό δέρμα, για να το πω έτσι, εντός εικόνα, αλλά και πολλοί συνηθισμένο ήταν σε περιπτώσεις ε, χωρισμών και σε αμυγός ε, γερμανικέ οικογένειε. Άρα, εγώ εργάζομαι εδώ και χρόνια με τι γυναίκε. Ξέρω πολύ καλά ότι δεν είναι ένα πρόσφατο φαινόμενο. Πώ θα το ξεκαθαρίσουμε αυτό, λοιπόν, ότι είναι ψευδή είδηση αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Πριν δώσω το λόγο για μια ακόμη φορά στους δύο προσκεκλημένους μας. Α, κύριε Άντερσον, θέλετε κι εσείς να κάνετε μια ερώτηση. Παρακαλώ, υπάρχει κάποιο άλλο. Να σηκώσετε τα χέρια σας τώρα, παρακαλώ. Ωραία, κύριε Άντρισον. Ναι, σύντομα σε σχέση με όσα έχουν ε, ήδη αναφερθεί στο δεύτερο τη βία σε βάρος των γυναικών ε, για τη ε, Σουηδία. Αν κατάλαβα καλά, είπατε ότι η βία μπορεί να είναι πιο υψηλή στη Σουηδία από τις χώρες των Βαλκανίων. Αυτό που βασίζεται, σε τι στοιχεία βασίζεται, αν κατάλαβα καλά από αυτά που είπατε και πράγματι πάντα υπήρχε βία σε βάρος των γυναικών στη στο δυτικό κόσμο. Ε, όμως μέχρι τώρα δεν ήταν ε, τόσο πολύ προβεβλημένο, δεν ήταν σημαντική διάταξη. Ε, δεν δινόταν ίσως ιδέουσα προσοχή. Εκτός μικροφώνου κάποιο σχόλιο. Και μια τελευταία λέξη να μα πείτε για τη βία στο Λοιπόν, ε, πριν δώσω το λόγο, λέει πρόεδρο, ε, στου προσκεκλημένου μα, θέλω να εκφράσω ένα πολύ μεγάλο έπαινο ότι και από, ε, σε επίπεδο Δήμων, σε επίπεδο κρατών, ε, σε ε, επίπεδο επίσης ευρωπαϊκό, ακούω τα καλύτερα για το έργο του ΕΓΚΕ, του Ινστιτούτου για την Ισότητα των είναι με μια πάρα πολύ σημαντική βοήθεια και υποστήριξη για πολλές χώρες που δεν μπορούν να συλλέξουν αυτά τα δεδομένα. Είναι ένα ευρωπαϊκό καθήκον δηλαδή αυτό το οποίο κάνετε, αλλά παίρνει διαστάσεις εθνικές και δημοτικές ε, δηλαδή ε, βοηθάτε και πράγματα τα οποία μένουν κρυφά ενδεχομένως σε εθνικό επίπεδο να δουν το φως, ε, να προβληθούν προς τα έξω. Επομένως, πραγματικά είναι αξιέπαινη η προσπάθεια του ΕΙΚΕ. Και το ερώτημά μου έχει να κάνει πιο πολύ με το μελλοντικό σας έργο και η ερώτηση μου είναι τι σας χρειάζεται, τι χρειάζεστε ακόμη. Τι ανάγκες έχετε για το μέλλον. Ποιος θέλει πρώτος το λόγο. Ανάποδα αυτή τη φορά. Κυρία Μπάρ θα ξεκινήσει. Thank you so much. Thank you for lot of very interesting. Σας ευχαριστώ. Πολλές και ενδιαφέρουσες ήταν οι ερωτήσεις σας. Ίσως ε, θα πρέπει να μιλήσουμε για το mainstreaming και την εργασία αυτού του οργανισμού. Θα ήθελα να σας πω ότι πρόκειται για πολύτιμες ε, και ε, πληροφορίες και πάρα πολλές πληροφορίες. Παρακαλώ χρησιμοποιήστε τες. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να είμαστε σε επαφή με το ΕΙΓΕ και τα απορίσματά του. Στις 15 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει ο νέος δείκτης ισότητας ε, των φύλων εδώ στις Βρυξέλλες. Φέτος ε, θα εστιάσει στην ισορροπία μεταξύ οικογενειακής και εργασιακής ζωής. Είμαι βεβαία ότι πάλι θα φέρω μαζί πολλές καινούργιες γνώσεις για αυτό το θέμα. Ε, reliability. Όσον αφορά την αξιοπιστία των δεδομένων και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων, ξέρετε για μένα ήταν πραγματικά εντυπωσιακό ότι ακόμα και όσον αφορά τις στατιστικές περί ε, μισθών, περί αμοιβών και υπάρχουν χώρες που ε, θεωρούν αυτά τα στοιχεία προσωπικά δεδομένα. Και άρα δεν μπορούν να τα δημοσιεύουν. Είναι δηλαδή τελείως διαφορετική κατάσταση σε κάθε χώρα. Ακόμα και όσον αφορά τους ορισμούς, έχετε πολύ δίκιο ότι οι ορισμοί κάποιες φορές διαφέρουν πολύ. Κυρίως στον τομέα της βίας. Ε, η συλλογή των δεδομένων ε, στην ε, Eurostat και η σύγκριση μεταξύ τους βασίζεται στην ίδια μεθοδολογία. Όσον αφορά λοιπόν τα δεδομένα της Eurostat, αυτά είναι πραγματικά αξιόπιστα. Είμαι πεπισμένη ότι τα στοιχεία που προέρχονται από τη Eurostat λοιπόν ε, είναι αξιόπιστα. Τώρα, τα καλά νέα είναι ότι οι ευρωπαϊκές στατιστικές έχουν εμπλουτιστεί με έναν από τους καλύτερους στατιστικολόγους του ΑΕΓΕ που μας βοηθά να ξεκινήσουμε τις στατιστικές με βάση το φύλλο σε πολλούς τομείς. Έχουμε λοιπόν πολλούς ε, τομείς όπου υπάρχουν στατιστικές με βάση το φύλλο όσον αφορά την απασχόληση, τον χρόνο, τα χρήματα, Υπάρχουν πολλά πολύτιμα δεδομένα. Ε, as far as ε, regional data, please ε, open the... Όσον αφορά την περιφερειακή εργασία, αν δείτε στη σελίδα του ΕΓΕ θα δείτε μια μελέτη που έχει εκπονηθεί για, για το φύλλο και το πώς αυτό εντάσσεται στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό διαπιστώνεται ότι όσον αφορά τα διευθυντικά ταμεία μόνο το 1% αυτών των κονδυλίων έχει στόχο προγράμματα που αφορούν το φύλλο και την ισότητα των φύλων. Για το ψηφιακό, ε, την ψηφιακή εποχή, ξέρω πως η ΑΕΚΕ έχει εγκύψει το θέμα. Βέβαια δεν είμαστε ειδικοί επαΐοντες. Περισσότερες φορές έχουμε πιο πολλά ερωτήματα από ό,τι απαντήσεις. Αλλά πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο πραγματικά είναι πρώτη προτεραιότητα της εργασίας του ΑΕΚΕ. Επιτρέψατε μου επίσης να πω κάτι όσον αφορά τις ψευδείς ειδήσει. Έχω την εντύπωση, την αίσθηση πως δεν είναι θέμα του ΕΙΓΕ να καταπολεμήσει τις ψευδείς ειδήσει. Ε, προσπαθούμε να σχηματίζουμε και να δίνουμε μία αξιόπιστη εικόνα για την ισότητα ή την ανισότητα. Υπάρχουν πολύ σοβαρές πηγές για τα δεδομένα όσον αφορά τις ε, ανισότητες, τις ανισότητες ε, την βία Κάποιες φορές μπορούμε να πιέσουμε ώστε να επαναληφθεί ή να ελεγχθεί μία μελέτη. Ε, χρειάζεται οπωσδήποτε να γίνει μία μελέτη για τη βία στην Ευρώπη, ε, γιατί πρέπει να έχουμε μια πραγματική εικόνα για το τι συμβαίνει. Εμείς είμαστε τα μάτια σας και τα αυτιά σας στο ειδικό φόρουμ του ΑΕΓΕ, αλλά σας παρακαλούμε να κάνετε κι εσείς ό,τι μπορείτε, ώστε να υπάρξει καλή συνεργασία με το οργανισμό αυτό, γιατί από καιρού εις καιρό φαίνεται να γίνονται απόπειρες για συγχώνευση αυτού του οργανισμού με άλλα οργανισμούς. Και έχω την αίσθηση πως ήταν αυτό μεγάλη απώλεια όσον αφορά τον αγώνα υπέρ της ισότητας των φύλων. Thanks. I will... Ο κύριος Γκούσταυσον, εγώ θα κάνω αυτό που υποσχέθηκα και τώρα θα μιλήσω σου ειδικά. Mm. Ευχαριστώ. Η Edit ε, ήδη απάντησε σε κάποιες από τις ερωτήσεις, επομένως εγώ θα προσθέσω κάποια πράγματα. Αν μας διέφυγε κάτι μπορείτε να μας ε, το υπενθυμίσετε. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθείτε είναι ότι η Edit και εγώ δεν εργαζόμαστε στο Ινστιτούτο αυτό αυτό. είμαστε στο Φόρουμ των Εμπειρογνωμόνων, επομένως δεν έχουμε απαντήσει για όλες τις ερωτήσεις. Γίνεται πάρα πολλή δουλειά για την εκπόνηση εκθέσεων, για τη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών και πραγματικά πιστέψαμε ότι θα μπορούσαμε να σας βοηθήσουμε αν σας ενδιαφέρει να διαδώσετε αυτές τις πληροφορίες ή αν ενδιαφέρεστε για περαιτέρω διάδοση αυτών των πληροφορών μπορούμε να σας βοηθήσουμε ή μπορεί να σας βοηθήσει η γραμματεία μας. Διορθώστε με αν κάνω λάθος ε, edit, αλλά αλλά υπάρχει μια πολύ πρόσφατη έκθεση για τη διαδικτυακή βία κατά των νέων κοριτσιών. Ε, το επιβεβαιώνει έτσι και είναι πολύ σημαντικό σημείο αυτό διότι αναφέρθηκε. Βλέπετε εκεί ότι υπάρχει σχεδόν κλιμάκωση της διαδικτυακής βίας και τα θύματα είναι κυρίως ε, νέα κορίτσια. Πρόκειται λοιπόν για κάτι το οποίο θα πρέπει να διαρευνήσουμε περαιτέρω και να κάνουμε περισσότερη δουλειά. Να δούμε τι ακριβώς είναι αυτή η διαδικτυακή βία, διότι πολύ δύσκολα μπορεί να δει κανείς μια τέτοια μορφή βία, αν αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Πολλοί από εσά ε, ανέφεραν τη Eurostat ε, και το πόσο σημαντικό είναι να πιέσουμε και εμείς να έχουμε περισσότερα στατιστικά στοιχεία, πιο αξιόπιστα στοιχεία, ώστε να μπορούμε να λαμβάνουμε τις κατάλληλες πληροφορίες. Ε, το κάθε κράτος μέλος όμως έχει διαφορετικό τρόπο ε, διαχείρισης των δεδομένων. Θα πρέπει να υπάρχει κάποιος τρόπος να συντονίσουμε τα στατιστικά στοιχεία για να μπορούμε να έχουμε συγκρίσιμα στοιχεία και ο ρόλος της Eurostat είναι κομβικός εδώ, διότι αυτή μπορεί να μας δώσει τέτοια στοιχεία. Η πρόεδρος επίσης είπε ότι οι πληροφορίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, διότι δεν είναι μόνο ε, θέμα ε, διαβίβασης των στατιστικών στοιχείων στη Eurostat. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τις πληροφορίες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Τώρα, τα fake news, οι ψευδείς ειδήσει, πολύ σημαντικό θέμα και αυτό. Μπορεί να με κατηγορήσει κανείς ε, για αφέλεια ίσως, αλλά είναι τεράστιο το πρόβλημα με τα fake news, αλλά δεν πιστεύω ότι θα μπορέσουν να κερδίσουν τη μάχη τελικά οι ψευδείς ειδήσει. Διότι όλοι εμείς είμαστε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και ο ΑΕΓΕ, ο οργανισμός είναι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λέμε, κάνουμε πράγματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αυτό αποτελεί αντίβαρο ε, στα ψευδείς ειδήσει. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν πάρα πολλές ψευδείς ειδήσει, υπάρχουν τομείς ε, οι οποίοι έχουν ε, διαχειριστεί κάπως καλύτερα αυτή την επίθεση και κάπως έχει αλλάξει ε, η κατάσταση σε σχέση με νωρίτερα. Νομίζω λοιπόν ότι είμαστε όλοι υπεύθυνοι να εξασφαλίσουμε ότι ό,τι δημοσιεύουμε είναι σωστό, αληθές, ε, να μπορούμε επίσης να απαντήσουμε σε ψευδείς ειδήσει με τα όσα ε, γράφουμε στο διαδίκτυο. Το γεγονός ότι οι ψευδείς ειδήσει έχουν κάποια επιρροή απορρέει ακριβώς από το γεγονός ότι αυτοί που τη διαβάζουν την είδωση ε, την πιστεύουν. Ε, αλλά όπως είπα μπορεί να είναι και δική μου αφέλεια αυτή. Ευχαριστώ. <laughs> Ναι. Σα ευχαριστώ πολύ. Και σε σχέση και με τα κοινωνικά δίκτυα μας δώσατε πάρα πολύ ε, καλές ε, πληροφορίες, μας δώσατε απλές ε, απαντήσεις και πραγματικά νομίζω ότι στην κοινωνία που ζούμε ε, πρέπει να υπάρχει το Ινστιτούτο σας ε, γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αυτά τα δεδομένα ώστε να μπορέσουμε να εργαστούμε έχοντας εμπιστοσύνη, έχοντας αξιόπιστα στοιχεία και Υπάρχει ομάδα εργασίας με μέλη από κάθε πολιτική ομάδα της ε, Επιτροπής μας και θα απασχοληθούμε με, θα ασχοληθούμε με το έργο του ΕΙΓΕ και ελπίζω να μπορέσουμε να αναπτύξουμε την καλύτερη δυνατή συνεργασία για να μπορέσουμε να αντιλήσουμε το μέγιστο δυνατόφελος από το Ε.Γ.Ε. και να δούμε τι άλλα στοιχεία μπορείτε να ε, παραγάγετε. Σίγουρα θα προκύψουν και νέα ερωτήματα. Ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό αυτό που είπατε. Σίγουρα έχει αναπτυχθεί η κοινωνία περισσότερο και ανακύπτουν συνεχώς νέα ζητήματα, νέα ερωτήματα ε, και τα δεδομένα τα οποία έχουμε, ναι, είναι σημαντικά, αλλά πολλές φορές δεν αποκρίνονται στην πραγματικότητα, δεν είναι επικαιροποιημένα για να μπορούν να μας βοηθήσουν τα πλούτα που έχουμε άμεσα να αντιμετωπίσουμε. Και επίσης έχουμε και την 15η ε, Οκτωβρίου για τον ε, δίκτυ της ε, ισότητας των Φίλων και να δούμε τι θα προκύψει γιατί σίγουρα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα για την Επιτροπή μας ε, και σίγουρα ε, ε, το έργο το οποίο κάνετε είναι πάρα πολύ σημαντικό και μπορείτε να βοηθήσετε όχι μόνο εμάς εδώ αλλά γενικώ τη χάρη πολιτική. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο σας και σας ευχαριστούμε θερμά εξ ονόματο της Επιτροπής μας για την επίσκεψή σας εδώ.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 Να προχωρήσουμε. Όσοι δεν έχουν λόγο να βρίσκονται για αυτό το σημείο να αποχωρήσουν και όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν να καθίσουν παρακαλώ. Περνάμε λοιπόν ε, στο επόμενο σημείο της ε, ημερήσιας ε, διάταξης το οποίο είναι Γενικός Υπερπολισμός Ευρωπαϊκής το Οικονομικού έτος 2020, όλα τα τμήματα. Η Φράνσις Φιτζέλντιν Σογήτρα, παρακαλώ έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχάς να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία να σας ευχαριστήσω για την ε, πολύ καλή συνεργασία και την επικοδομητική μας ε, ε, πρόοδο. Έχουμε κάνει πρόοδο με τους διάφορους εκπροσώπους των ομάδων και αναμένονται θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε την επόμενη εβδομάδα τη Δευτέρα. Από ό,τι έχω καταλάβει αυτό είναι το σχέδιο. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω όλους όσους πέβαλαν τροπολογίες οι περισσότερες από αυτές προσπαθούσαν περισσότερο να απτύξουν και να βελτιώσουν το κείμενο, να αποφύγουν την επικάλυψη και να επιφέρουν σαφήνεια στα αιτήματά μας. Η έκθεση αυτή είναι καλό προηγούμενο για το πώς εργαζόμαστε στην Επιτροπή αυτή όσον αφορά τη συνεργασία και ελπίζω πως οι εμπειρίες ε, των συναδέλφων είναι το ίδιο επικοδομητικές με τις δικές μου, γιατί πιστεύω πως αν συνεργαστούμε εντός της Επιτροπής με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα μπορέσουμε να οθήσουμε το δυναμικό των γυναικών στην Ένωση και θα στρίξουμε τις γυναίκες αντιμετωπίζοντας τα κύρια ζητήματα που προβληματίζουν τα μέλη αυτής της Επιτροπής. Να πω επίσης πως και η Γραμματεία έκανε πολύ καλή δουλειά με το κείμενο, με τις τροπολογίες και θέλω να τους ευχαριστήσω όλους ιδιαίτερος. Δεν το βλέπουμε αυτή τη δουλειά. Είναι ε, ε, υποστήριξη όμως. Ευχαριστώ λοιπόν για την στήριξη αυτή και όπως είπα νομίζω θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε την επόμενη Δευτέρα το απόγευμα. Και εγώ σας ευχαριστώ Φράνσις Φιτζέραλντ. Η Μαρία. Μάλιστα. Ήθελα να ευχαριστήσω για, την, ε, για το έργο που έγινε και η γραμματεία συνέβαλε με τις ε, τροπολογίες ε, και θέλω να σας ευχαριστήσω και σας προσωπικά. Πέντε χρόνια εργάζομαι στο Ευρωκοινοβούλιο και είχα την ευκαιρία να συναντήσω πολλές γυναίκες, αλλά πραγματικά ε, διαπιστώνω ότι εσείς έχετε την αίσθηση του καθήκοντος και σε προσωπικό επίπεδο είστε εξαιρετικός άνθρωπος για την ε, αγώνα υπέρ των γυναικών. Δεν μπορώ να προσθέσω πια τίποτα παρά να σας ευχαριστήσω για, ε, για το έργο σας. Ευχαριστήσαμε και την γραμματεία, αλλά κυρίως εσάς πρέπει να ευχαριστήσω και ελπίζω να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με τόσο επικοδομητικό τρόπο. Είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Και πάλι ευχαριστώ. Ε, πολύ ευχάριστο να ακούμε τέτοια κοπλιμέντα και κυρίως ότι λειτουργεί αγαστά η συνεργασία. Αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Και... was our shadow, couldn't Μονίκα Βανά που ήταν σκιώδης δεν μπορούσε να είναι παρούσα. Ήθελε και εκείνη να είναι εδώ και να ευχαριστήσει την κυρία Φιτζέραλτ, την εισηγήτρια, για την εργασία της. Ε, και η Μονίκ Βανά ε, εργάστηκε πολύ για την ένταξη του θέματος των φίλων στον προπολογισμό και ήθελε να κάνει κάποιες δηλώσεις για αυτό τον προπολογισμό. Ήδη με την αρχή αυτής της αιτίας ε, φάνηκε να υπάρχουν κάποιες θετικές αλλαγές. 70 εκατομμύρια ευρώ θα δαπανηθούν για το φύλλο και για την ανθρώπινη ε, ανάπτυξη και χρηματοδότηση για την προώθηση του προγράμματος για τα φύλλα και αυτό θα φανεί και στην ενδιάμεση αναθεώρηση του PDP. Θέλαμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι σωστό να επιμείνουμε γιατί ο προπολογισμό ποτέ δεν είναι ουδέτερος όσον αφορά τα φύλλα. Αντίθετα, η κατανομή του είναι αυτή που επηρεάζει την ισότητα, την ανισότητα των φύλων. Έχουμε επιτύχει πολλά ήδη, αλλά πρέπει να γίνουν και άλλα πολλά, να γίνονται καλύτερες αναλύσεις, ώστε να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να δαπονηθούν τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογούμενων και να μην επιβαρύνονται οι γυναίκες. Τα σημεία που πραγματικά θέλαμε να πούμε στην Επιτροπή Προϋπολογισμού είναι ότι η ισότητα των φύλων θα πρέπει να ενταχθεί σε όλες τις πολιτικές και στις αποφάσεις προϋπολογισμού, όχι μόνο σε αυτές που προφανώς αφορούν το φύλο. Δεύτερη παρατήρηση. Οι ευρωπαϊκές επενδύσεις θα πρέπει να θαρρύνουν μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Τρίτη παρατήρηση. Οποτεδήποτε ε, ανανεώνουμε την έκκλησή μας για προώθηση των γυναικών και των κοινωνικών τους δικαιωμάτων, ιδιαίτερα όσον αφορά τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Και τέλος, τέταρτη παρατήρηση. πιστώνουμε ότι μειώθηκαν ε, ε, τα χρήματα όσον αφορά την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και θα θέλαμε να ξαναυξηθεί το κονδύλι θέλω να σας πω ότι το gender budgeting ε, ε, στην ε, Αυστρία είναι σταματικά κατοχυρωμένο. Θα το έλεγε και η Μόνικα Βάνα αν ήταν εδώ. Και υπάρχει σίγουρα μεγάλη επιρροή και σε ό,τι αφορά την απασχόληση ανδρών και γυναικών, άρα δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω Θέλει κάποιος άλλος το λόγο, αν όχι να δώσω ξανά το λόγο στην εισηγήτρια. Κανείς δεν θέλει το λόγο από ό,τι βλέπω. Άρα δεν ξέρω αν θέλετε κύριε Φιτσέλαλτ να κάνετε έτσι μια επισκόπηση. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Να σας ευχαριστήσω και για την υποστήριξη. Να ευχαριστήσω και το προσωπικό που εργάζεται μαζί μου. Νομίζω ότι σημαντικά πράγματα θέλουμε να έχουμε τον προπολογισμό. Και σίγουρα εξίσου σημαντική είναι και η παρακολούθηση τη υλοποίηση του προπολογισμού. Το είπε και τελευταία ομιλήτρια. Με το gender budgeting ε, μπορούμε πραγματικά να παρακολουθούμε τι γίνεται στην πράξη. Άλλο η θεωρία και άλλο η πράξη. Το ότι πραγματικά μπορεί να δει κανεί ε, ότι κάθε χρόνο έχουμε επιτυχίες και για τα επόμενα πέντε χρόνια πρέπει να το φροντίσουμε να μην μένουμε στα θεωρητικά, στις θεωρητικές δεσμεύσεις, αλλά στην πράξη να βλέπουμε ότι επηρεάζεται η χρηματοδότηση ε, μέσω διαφόρων ταμείων και να το βλέπουμε παντού, όχι σε λίγους τομείς μόνο. Διότι πραγματικά οι επιπτώσεις ε, είναι πολύ σημαντικές. Είπατε κι εσείς ε, για την απασχόληση. Επίσης, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παντού έχει σημασία. Ευχαριστώ πολύ και σίγουρα η παρακολούθηση θα είναι κάτι σημαντικό Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ και έτσι, για να επαναλάβω αυτό που είπε η Φράνσις ε, η ψηφοφορία στην Επιτροπή λαμβάνει χώρα ε, στις 30 Σεπτεμβρίου, ε, το απόγευμα στις 5 τη Δευτέρα. Ε, δεν ξέρω ακριβώς τι θα γίνει με τις ακροάσεις. Ε, ε, καλό θα ήταν να είμαστε όλοι παρόντες. θα ψηφίσουμε λοιπόν στις 5 στις 30 Σεπτεμβρίου και η ψηφοφορία στην Επιτροπή Προπολογισμών θα λάβει χώρα στις 14 Οκτωβρίου. Και τώρα έρχομαι στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Βλέπετε ότι προχώρησαν πάρα πολύ γρήγορα σήμερα στο σημείο 7 διάφορα. Υπάρχει κάτι υπό τα διάφορα. Ούτως ή άλλως θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα και φαντάζομαι ότι όλοι είστε απασχολημένοι με την προετοιμασία των ακροάσεων για να εκφράσουμε τις απόψεις μας καθαρά και δυνατά. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ε, παρισταμένους. Να ευχαριστήσω βέβαια και τους διερμηνείς. Σας εύχομαι καλό απόγευμα και μια καλή εβδομάδα.